παντός. Διαφορετικά, ε, ο Αλέξης Κινάς θα έχει το χατοφυλάκιό του, αλλά έχει όμως Αμερικανούς και τους Κινέζους που θα αποφασίζουν ε, αντί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ανταποκριθούμε κατάλληλα στις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Κέλλερ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί υποψήφοι επίτροποι, σήμερα ε, θέλετε να εκλεγείτε για να καθοδηγήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ένωση που προέκυψε μέσα από ένα αγώνα για τη δημοκρατία, την ειρήνη. Ένα ε, πραγματικά εντυπωσιακό εγχείρημα. Τώρα, αν δούμε ε, αν στρέψουμε το βλέμμα μας, θα δούμε ότι πολλοί άνθρωποι πνίγονται στα σύνορά μας. Ε, πολλές γυναίκες δολοφονούνται και σε και κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποστρέφουν το βλέμμα από το κράτος δικαίου, από την ελευθερία, κάτι και όλα αυτά για τα οποία εργάστηκαν και πάλεψαν τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι. Μία Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική κρίση, η οποία βλέπει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή το, της αυτής της αλλά και της μελλοντική. Είναι όμως και μία ένωση με πολλές δυνατότητες να είναι στεχμή του δόρατος ε, για την προστασία του κλίματος. Ε, μία ήπειρος ε, η οποία αγωνίζεται για τις αξίες της, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είτε στην Ευρώπη είτε και γενικότερα στον κόσμο. Σήμερα λοιπόν το διακύβευμα είναι το εξή. Κατά πόσον η Νέα Επιτροπή εσείς θα είστε έτοιμοι για να εκμεταλλευτείτε όλο αυτό το δυναμικό, να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις σε επίπεδο περιβάλλοντος, σε δημοκρατία και σε πολλά άλλα επίπεδα. Αυτά που είναι σήμερα μάστιγα για την Ευρώπη. Αυτό όμως απαιτεί θάρρος. Και κατά τη διάρκεια των ακροάσεων ακούσαμε κάποιους από εσά ε, να είναι στρατευμένοι, αλλά δεν ισχύει για όλους, ούτε για όλα τα θέματα. Παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα προσφέρει ένα φιλόδοξο περιβαλλοντικό πρόγραμμα αν δεν υπάρχει βούληση να αλλάξει η γεωργική και η εμπορική πολιτική. Εγώ σας λέω, δεν θα τα καταφέρετε. Ε, δεν αρκεί αυτό που λέτε. Χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο, μια πιο φιλόδοξη μερίσια διάταξη. Χωρίς βαθιά αλλαγή της ε, γεωργική πολιτική και τη εμπορική πολιτική, ε, το κλίμα θα υποφέρει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει πια χρόνος για να αλλάξουν όλα αυτά. Και επιτρέψτε μου να σας επισημάνω και κάποια άλλα προβλήματα. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση το γεγονός ότι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ε, πληροφορικής στην Ευρώπη έχει έναν ε, δικό της άνθρωπο, τον επίτροπο που θα είναι αρμόδιος για την εσωτερική αγορά. Ε, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε βέβαια αυτά τα οποία έχει αναλάβει ο Επίτροπος να κάνει για να ελαχιστοποιήσει τη σύγκρουση συμφερόντων. Πιστεύουμε όμως ότι η σύγκρουση συμφερόντων είναι εγγενής, ε, είναι συνειφασμένη στο χαρτοφυλάκιό του. Ε, και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ψηφιακή αγορά θα έπρεπε να έχει αφαιρεθεί από το χαρτοφυλάκιό του. Εμείς ως πράσινοι δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί αυτό θέτει σε κίνδυνο τη φήμη μας ως ευρωπαϊκή θεσμή. Άλλο μεγάλο πρόβλημα αφορά τον Επίτροπο από την Ουγγαρία που μας τον έστειλε με τους θερμού του χαιρετισμού ο κύριο Όρμπαν. Πώ είναι δυνατόν κάποιο ο οποίο εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που μονίμω υπονομεύει και παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και τι αξίε, ε, πώ μπορεί ένα τέτοιο άνθρωπο ε, να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λένε οι υπόλοιποι να εφαρμόζουν το κράτο δικαίου. Ε, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι τουλάχιστον κοινικό. Και πιστεύω ότι οτιδήποτε αφορά τα ευρωπαϊκά ε, ιδεώδη Οτιδήποτε λοιπόν αφορά αυτά τα ιδεώδη σημαίνει ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στην δημοκρατία, την ελευθερία. Ε, για μας αυτό σημαίνει Ευρώπη. Και τι μπορούμε να πούμε σε εκείνες τις χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή θέλουν να αλλάξουν την ε, πολιτική τους. Άλλαξαν ακόμα και το όνομά τους. Ξέρετε τι σου λέμε δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν έχει καμία σημασία, δεν εισακούει τη φωνή του, δεν έχουν σημασία οι προδοξίε του. Λάθο αυτά που έγιναν σε αυτό το τομέα πρόσφατα, α μην ξανακάνουμε κι άλλα λάθη. Κυρία Πρόεδρε, αυτά τα θέματα δεν σταματήσαμε να τα θέτουμε επιτάπητος. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά για αυτούς ακριβώς λόγους εμείς δεν θα σας στηρίξουμε. Είμαστε βέβαια πρόθυμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσουμε την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, για να προαχθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οποτεδήποτε εσείς οι συνάδελφοί σας αναλαμβάνετε πρωτοβουλίε σε αυτόν τον τομέα ή σε αυτού του τομείς, θα συνεργαστούμε συνεργαστούμε μαζί σας. Ε, θα βρείτε σε μας έναν επικοδομητικό συνεργάτη, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα ασκούμε επίσης ε, κριτική. Μπορείτε να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, πρέπει να δράσουμε. Το κλίμα δεν μπορεί να περιμένει πια ούτε η ευικία και η ανισότητα. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η Επιτροπή θα μας εκπλήξει με πολλούς θετικούς τρόπους και ελπίζουμε να μας δώσετε ήδη από σήμερα ένα καλό δείγμα. Καλή τύχη. Ευχαριστώ για το ID. Ο κύριος Μπαρντέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Βάντερ Λάιν στη συζήτηση ε, αριστερή και δεξιά δημιούργησαν ε, την εντύπωση διαφωνίας στις εκλογές για την κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα μέσω συγκερασμού συμφερόντων θα εκλέξετε μία ε, κομισιόν η οποία συνεχίζει την προηγούμενη. Ε, λοιπόν, βλέπουμε αλλαγή θέσεων ε, απλώ στα χαρτοφυλάκια θα κάνει καλό. Ένα καλό επίτροπο είναι εκείνο ή εκείνη που μπορεί ε, να κινηθεί εντό των κανονισμών και των διαδικασιών που το μυστικό όμω αυτόν το κατάει οι Βρυξέλλε. Οι πολιτικέ δυνάμει περάσσονται τα συμφέροντα των εθνών και των κρατών έπρεπε να σωθήσουν να δείτε αλλιώ ε, ότι χρησιμοποιείται την, ε, την προσέγγιση που είναι απερχαιωμένη. Ε, Αθέμητο ανταγωνισμό, αποσπασμένο εργαζόμενο, φιλελευθερωποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, ο, Ομοσπονδιακή Ευρώπη και χαλά, χαλαρή προσέγγιση στη μετανάστευση. Λοιπόν, τελικά τεχνοκρατικά θα κινηθείτε χωρί σύνορα και χωρί όπλα με αυτά που προτείνετε. Λοιπόν, δίνετε, έχουν για την προστασία της, ε, για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και θα γίνει η πρόθεση του τρόπου ευρωπαϊκής ζωής από κάποιο σοσιαλιστή. και θα είναι ένας επίτροπος για την πρόθεση της μετανάστευσης τελικά. Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι θα παίξει το ρόλο της, δηλαδή να προσπαθεί να πνίξει την ελευθερία και την ιστορική συνέχεια των εθνών της Ευρώπης. Το Brexit είναι ευκαιρία για το Συμβούλιο να ξανεξετάσει τη συνθήκη και να έχουμε πιο δίκαιη Ευρώπη των εθνών, πιο προστατευτική πιο δημοκρατική. Juncker, von der Leyen, ένα παιχνίδι αλλαγή θέσεων, ένα παιχνίδι ε, που αλλάζουν οι καρέκλες, αλλά δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα. Συνάδελφε Φίτο. Εσεί έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μα θέση σήμερα ξεκινά από ένα στοιχείο. Τη συζήτηση δηλαδή που ακούσαμε και από τόσα προγράμματα και ενδείξεις, υποδείξεις που προέκυψαν από αυτήν ε, την συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα σημείο κίνησης το οποίο αγνοείται. Είναι η δουλειά της Επιτροπής Juncker. Είναι το πρώτο σημείο απόκλησης όπου εμείς είμαστε τελείως αρνητικοί ως προς την κρίση μας γιατί η Επιτροπή Juncker τα τελευταία πέντε χρόνια έκανε, ήταν τόσο αργή ε, στην πολιτική της για την εξέβρεση λύσεων που ακόμα και εκεί που τις βρήκε ε, τις λύσεις τα προβλήματα είχαν τελικά αλλάξει μέχρι ότου βρεθούν οι λύσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε Ποια είναι το πολιτικό ζήτημα. Ε, ε χτες ε, έγινε πρόταση, ας πούμε, ένα κείμενο πρόταση από πλευράς Γερμανίας και Γαλλίας και στην ουσία αφορά ε, την θέση και τη στάση της, Ευρω... της Επιτροπής Juncker που έφερε σε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Και εδώ προστίθεται άλλο ένα ζήτημα που είναι το ίδιο σημαντικό. Οι διαφορές που χαρακτήρισαν τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στις τελευταίες μέρες και του τελευταίους μήνες ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία Γερμανία και όχι για ε, ίσονο σημασία θέματα. Το να έχουμε διαφορετική και ε, επικριτική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ δεν είναι το ίδιο στο εσωτερικό αυτών των θεσμών. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτέ μα τι θέσει, να δούμε τι θέλουμε. Ε, σε αυτά τα πράγματα θέλουμε ξεκάθαρε θέσει και έπειτα υπάρχουν και θέματα. Βεβαίω η ομιλία τη Προέδρου τη Επιτροπή και το πρόγραμμα το οποίο είναι στραμμένο προ το μέλλον και που στόχο έχει να λύσει όλα τα σημαντικά θέματα που έχουμε επιτάπητος, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Ναι, λέει Just a Transition Fund. Πώς το θέμα της μείωσης των εκπομπών. Να το βάλουμε όχι σε μια λογική ε, περιβαλλοντική περιβαλλοντικού εξεμισμού, αλλά να βρούμε κάποιες σταθερές. Το 9% των εκπομπών παγκοσμίω προαγράγεται στην Ευρώπη πέρα από το 40% δηλαδή αφορά πάνω από το 40% αφορά τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Και ποια είναι η πολιτική μας βιομηχανική πολιτική, ποια είναι η απάντησή μας στον κόσμο της εργασίας, τις επιλογές που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, το πρόβλημα του ευρωπαϊκού προπολογισμού για τα επόμενα 7 χρόνια. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα, ναι. Πράσινο σύμφωνο, πολιτική συνοχή, πολιτική γεωργία κτλ. Πώ θα γίνει αυτό, πώ θα λυθεί ο γόρδιο δεσμό του προπολογισμού προπολογισμού, ε, ε, ε, όπως επίσης το σπουδαίο θέμα του προπολογισμού, όπου μπορεί και ακόμα μια φορά να μπει η καθυστέρηση και οι μηχανισμοί ποινών για διάφορες χώρε. όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν με το άρθρο 7. Να βρούμε λύσεις, απαντήσεις για τις χώρες όπου ενεργοποιήθηκε αυτή η διαδικασία από πλευρά του κόσμου, γιατί στις χώρες αυτές οι εκλογές έδωσαν αντίθετη απάντηση στην δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίχθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Για αυτά τα ζητήματα λοιπόν χρειάζεται σαφήνεια. Επίσης θέλω τελευταίο να αγγίξω και το θέμα της μετανάστευση. Η δικιά σας έκκληση και αναφορά σα στη δραματική περίπτωση ε, των 39 ε, νεκρών μέσα σε ένα φορτηγό Βεβαίω μας κάνει να προβληματιστούμε. Αλλά αυτό σημαίνει αποτυχία γιατί στις, 29, ε, στις 21 Νοεμβρίου πνίγηκαν 77 μετανάστες και από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι σήμερα χάθηκαν χίλια άνθρωποι. Ποια είναι λοιπόν η πολιτική. Υποσχόμαστε περισσότερους πόρου μέσα στον ε, προπολογισμό για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και να στηρίξουμε τις αστυνομικέ δυνάμεις φύλαξη των συνόρων ή πραγματική και σοβαρή απάντηση και να δώσουμε ευθύνη σε όλους και να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα εκεί όπου ε, ξεκινούν οι μετανάστες, όχι στο σημείο άφηξής τους δηλαδή. Αυτά είναι προβλήματα που εμείς θέτουμε. Η ομάδα μας έχει διαφορετικοποιημένη θέση. Δεν είναι τίποτα το κρυφό. Είναι γνωστό πως έχουμε στο εσωτερικό μας ένα κόμμα το οποίο έχει και έναν επίτροπο. Δηλαδή η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Θα δούμε στα ζητήματα σημείο προ σημείο τις δράσεις και τις συνέπειες αυτών και από αυτόν θα συμβάλλουμε εκεί όπου η συμβολή μας θα είναι χρήσιμη. Εκεί όπου θα διαπιστώσουμε πως θα υπάρξει μια στρατηγική διαφορετική από τις δικές μας θέσεις, βεβαίως θα είμαστε αντίθετοι. Πολύ ωραία. Ο κύριος ε, Σιρντεβαν, παρακαλώ κύριε Σιρντεβαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Φοντελάιν. Έχουμε ένα πρόβλημα. Σήμερα, αλλά και τους ε, προηγούμενους μήνες, υποσχεθήκατε στους πάντες τα πάντα. Επενδύσεις, μέχρι και ένα δις, ε, ένα Green New Deal. Μιλάτε για πολλές και μεγάλες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, στην οικονομία, στην κοινωνία. Όμως, μέχρι τώρα δεν μπορέσατε να αντιμετωπίσετε την εξή αντίφαση. Όλα αυτά που υπόσχεστε, πώς θα τα κάνετε από τη στιγμή που θέλετε να επιβάλλετε περικοπές. Κυρία Φοντελάν, με το πολιτικό σας πρόγραμμα θα αποτύχετε αν δεν άρεται την πολιτική λιτότητα και δεν μπορούν τα κράτη πλέον να κάνουν επενδύσεις. Κύριε Φοντερ Λάιν, μπορεί να υπάρξει μια άλλη Ευρώπη, αλλά εμείς έχουμε διαφορετικά οράματα. Αλλιώς τα σκέφτεστε εσείς, αλλιώς εμείς, γιατί την ειρήνη δεν μπορεί κανείς να την επιτύχει με την στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής, αλλά αντίθετα επιβάλλοντας εμπάργο όπλων η κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να απορριθμίζει κανείς ε, τις εργασιακές ε, σχέσεις, αλλά επιβάλλοντας κοινωνικά πρότυπα, προστατεύοντας από τη φτώχεια. Η προστασία του κλίματος δεν χρειάζεται μεγαλεπίβολα λόγια, αλλά μια φιλόδοξη πολιτική έτσι ώστε η υπερθέρμανση του πλανήτη να κατέβει στο 1,5 βαθμούς ε, και οι εκπομπές να περιστούν μέχρι και 70%. Η φοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παραπέμποντας τον ΩΣΑ, αλλά επιβάλλοντας σωστούς επιχειρηματικούς φόρους και κλείνοντας τους φορολογικούς παραδείσους. Και τις ανθρώπινες ζωές δεν μπορεί κανείς να τις προστατεύσει με αυτή την στεγανοποίηση των εξωτερικών συνόρων, αλλά με μια κοινωνική αντιμετώπιση των ανθρώπων που μας χρειάζονται. Κυρίες και κύριοι, αγαπητή κυρία Φοντελάιν, εμείς εδώ ως αριστερά είμαστε μια ενωμένη δημιουργική αντιπολίτευση και σας το υπόσχομαι, κατά τα επόμενα πέντε έτη, κάθε μέρα θα είμαστε ε, θα σας παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων για να αλλάξει αυτή η πολιτική και να έχουμε μια διαφορετική Ευρώπη. Ευχαριστώ μη γεγραμμένη. Συνάδελφοι Μπεγκίν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Επίτροποι, συνάδελφοι, ε, Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε άμεσα με κυβέρνηση σαν Ευρώπη. Ήδη χάσαμε πάρα πολύ κόσμο και οι πολίτε μα ζητάνε απαντήσει που δεν μπορούν πλέον να περιμένουν. Δεν κρύβουμε ότι όχι όλη η ομάδα σα μα πείθει. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων είδαμε γιγάντιες συγκρούσεις συμφερόντων, ακούσαμε πάρα πολλά ναι, καδισταγμούς κλπ. Εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας περιμένουμε μόνο ναι, όχι, όχι. Ε, ναι, για την υποχρεωτική μετακατάσταση των μεταναστών. Ναι, στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητα. Ναι, στι ε, πράσινε επενδύσει. Ναι, στο Made in για να προστατεύσουμε τι επιχειρήσει μα. Χάρη σε αυτέ τι προτεραιότητε, εσεί τον Ιούλιο λάβατε την εμπιστοσύνη μα. Τώρα όμω οι πολίτε περιμένουν συγκεκριμένε δράσει. Υπάρχουν ε, εκατομμύρια εργαζόμενοι και κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργασία του λόγω τη υπερπαραγωγή του χάλιβα. Καλώ, α χρησιμοποιήσουμε το Just Transition Fund και για το χάλιβα, εκτό από τον άνθρακα. Οι αλλαγέ του κλίματο καταστρέφουν την Ιταλία. Να αντιδράσουμε αποκλείοντα από το Σύμφωνο Σταθερότητα του πόρου για την ανοικοδόμηση, για την πρόληψη, την υδρογεολογική. Κλείνοντα, το κίνημα πέντε αστέρων θα αξιολογήσει κάθε απόφαση και κάθε διάταξη επί τη ουσία. Λοιπόν, δεν θέλουμε να δώσουμε μία λευκό επιταγή. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Κάσπαρη, για 1,5 λεπτό έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον Ιούλιο ε, παρουσιάσατε ένα πιστικό πρόγραμμα, το πράξατε και σήμερα, ισορροπημένο το πρόγραμμά σας, σας συγχαίρω θερμά. Σήμερα λοιπόν, 30 ε, χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υπάρχει διαφθορά. Οι δημοσιογράφοι πολλές φορές φοβούνται για τη ζωή τους, μάλιστα και δολοφονούνται και σας είμαι ευγνώμων που το επισημάνατε. Πραγματικά πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν να επικρατήσει το κράτος δικαίου, η ελευθερία και η ειρήνη. Και για να τα πετύχετε αυτά σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ε, θίξατε το θέμα της ε, ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούσαμε πάρα πολλά χρόνια ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα εγγυούνται την ασφάλειά μας. Δυστυχώς όμως βιώνουμε ότι το κάνουν όλο και λιγότερο. Μόνοι μας πρέπει να φροντίσουμε για τη γειτονιά μας, μόνοι μας να διασφαλίσουμε στη γειτονιά μας να μην ε, υπάρχουν υπάρχουν ε, εκρήξεις εμφυλίων πολέμων, να μην δολοφονούνται εκατοντάδε ανθρώπων. εμεί πρέπει να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και αυτό είναι κάτι που θέλω να το προβάλλω. Πάω στο τρίτο, στην κλιματική αλλαγή. Σας είμαι ευγνώμων. Πράγματι χρειαζόμαστε το πράσινο σύμφωνο, αλλά το είπατε κι εσεί ότι δεν θα πρέπει να είναι μονόπλευρα πράσινο. Οι άνθρωποι το φοβούνται αυτό. Φοβούνται οι άνθρωποι που δουλεύουν στον Ιμάντα, στα εργοστάσια, στην Ήπεθρο, που νιώθουν απομονωμένοι. Ε, φοβούνται οι άνθρωποι που διρωτώνται τελικά πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η παραγωγή τροφίμων. Εσείς είπατε ότι πρέπει να επιδιώξουμε την βιωσιμότητα, να μην τρομάζουμε τους ανθρώπους, αλλά να τους πείσουμε ότι έχουμε πρόγραμμα, έχουμε προσανατολισμό, ιδέες για το μέλλον, τα είπατε όλα αυτά, σας είμαι ευγνώμων και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν είχαμε μια ανοιχτή, αισιόδοξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοιχτή και αισιόδοξη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό η κυρία Μποναφέ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Βόντερ Λόιεν, κύριε Επίτροπε, με τη σημερινή μα ψήφο ξεκινά μια νέα πορεία. Οι δεσμεύσει που εσεί αναφέρετε ε, παρουσιάσατε και τις οποίες στηρίζουμε θα πρέπει από αύριο να συγκεκριμενοποιηθούν σε μέτρα για να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας. Και στο υπόσχομαι θα είμαστε πιστοί αλλά πολύ απαιτητικοί στην επαλήθευση του προγράμματος. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις. Αντίθετα θα αυξήσουμε περισσότερο τη φιλοδοξία. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την εθνικιστικό άνεμο οι πολίτες δείξαν ότι έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία. Εμείς τώρα δεν θα πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Ε, εδώ, Επίτροπε Φοντερ Λάιεν, Επίτροπη, παραφράζοντας μια φράση ε, ενό διάσημου Ιταλού, εδώ φτιάχνουμε την Ευρώπη ή πεθαίνουμε. Έχουμε μια σειρά από προκλήσεις. Εγώ θέλω τρία πράγματα να τονίσω. Βιωσιμότητα για όλους, δικαιοσύνη κοινωνική. Πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε με ακρίβεια. Ε, ανάπτυξη για όλους που θα είναι βιώσιμη ε, περιβαλλοντικά. Για να ε, αναζωογονηθεί η οικονομική ζωή, να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης ε, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει νέα προσέγγιση στην οικονομική διακυβέρνηση που θα στοχεύει στη μεγέθυνση όχι μόνο με, οικονομικούς, ε, ε, με οικονομικές συνιστώσεις αλλά με κοινωνική ανάπτυξη επίση. και για να γίνει αυτό χρειάζεται και κατάλληλο προπολογισμό χωρί πόρου μπορεί να μείνουμε μόνο στα ωραία λόγια. Αυτά λοιπόν οι σοσιαλιστέ δημοκράτες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί, να δουλέψουμε χωρί φιδό και καθημερινά να αποδείξουμε στην Ένωση των των πολιτών που εκπροσωπούμε, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εγγύηση για το μέλλον όλων μας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Journay, for one and a half minutes. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ζουρνέ, για 1,5 σε λεπτοχώσετε, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ήδη συζητήσαμε αρκετά. Ε, πετύχατε πλειοψηφία εδώ στο ημικύκλιο, εδώ και κάποιου μήνε στι ακροάσει. Ακούσαμε στι ακροάσει όλου του επιτρόπου και εσεί γυρίσατε σε όλε τι ομάδε και τα επιχειρήματα συζητήθηκαν εκτενώ. Δεν θα υποβάλω συμπληρωματικέ ερωτήσει, αλλά προβώ σε ένα σχόλιο. Όπω όλο ο κόσμο εδώ, γνωρίζουμε ότι περνάμε μια στιγμή που είναι καμπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκω σε εκείνου που πιστεύουν ότι το ημικύκλιο δεν είναι αιώνιο και θα πρέπει να φροντίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, του θεσμού μα, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε το ευρωπαϊκό μας μοντέλο και το ευρωπαϊκό μας πολιτικό οικοδόμημα, το ευρωπαϊκό. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή μας η μελλοντική βγήκαν από μια δημοκρατική διαδικασία που αποτελείται από Ευρωπαίους πολιτικούς ανθρώπους και όχι επικεφαλής ε, διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε ενσάρκωση των δημοσίων πολιτικών και απευθύνομαι στο όλο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε ενσάρκωση των δημοσίων πολιτικών στα εντό τη Ευρώπη και στα μέσα να, να προβάλλεται η Ευρώπη και να δοθούν απαντήσει στι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών. Μα το είπαν ότι θέλουν αποτελεσματικότερη Ευρώπη στι εκλογέ. Μια Ευρώπη που αποδίδει, που μιλάει για προτεραιότητε που θέτει. Την ίδια παρέμβαση έκανε την προηγούμενη φορά στην ε, ε, πρώτη ψηφοφορία για την έγκρισή σας. δεν βλέπω τη θέση των πρασίνων σε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω, ε, μάλλον βλέπω πράσινο στίγμα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπω προοδευτική ε, κίνηση, αλλά δεν βλέπω επιχειρήματα. Κυρία Κέλλερ, ίσως να ξέρετε κάτι τα επιχειρήματα. Δεν βλέπω λόγους και επιχειρήματα για το αντίθετο. Σας ευχαριστώ για τις συζητήσεις, ευχαριστώ για τις προτεραιότητες και προφανώς θα υπερψηφίσουμε την Ευρωπαϊκή σας ε, Επιτροπή. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, να πω ότι προσπαθώ να είμαι ευέλικτη στον αυτό χρόνο, αλλά έχουμε ήδη 12 συναδέλφου στο Catch the Eye και θέλω να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα. Δεν λέω γιατί το έχετε το λόγο εσεί για ένα λεπτό, κύριε Σμιθ, το λέω για εσά, αλλά παρακαλώ να δώσετε το καλό παράδειγμα. Πάντα προσπαθώ να είμαι λακωνικό. Καλημέρα συνάδελφοι. Χαρά μου να είμαι εδώ Δόκτωρ Βόντεν το, εθνικό, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι το σωτικό μα πλαίσιο με το Brexit έχει χωματίσει τη σκέψη μα. Πρέπει όπω συναδέλφοι ότι ο κόσμο φαίνεται διαφορετικό αντιμετωπίζει κανεί την προοπτική χώρα σου να βγει παρά τη βούλησή σου από αυτή την οικογένεια των εθνών βλέπουμε την μεγάλη γενική εικόνα και σε λεπτομέρειε. Δόκτωρ Βοντερ Λάιν, χρειαζόμαστε νέο δυναμισμό στην Ευρώπη. Επί Μακρόν ήταν πολύ εύκολο να παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν κάτι που είναι στήρο, που δεν νοιάζεται για τίποτα και δεν έχει επαφή την πραγματικότητα. Ελπίζω εσεί και το νέο σα σώμα πράγματι να δώσετε νέα ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόεδρε, στην τελευταία μου ομιλία σε αυτό το σώμα είμαι ψήφιο για τι εκλογέ ε, για το Sterling στο Ηνωμένο Βασίλειο και, λοιπόν, και πρωτίστως ε, ίσως πρέπει να αποχωρήσω. Λοιπόν, η Ευρώπη ε, ευλόγησε μια γενιά να πρέπει να Υποστηρίξτε την Ευρώπη. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα στο οποίο συμμετέχετε. Μην το λησμονείτε. Είναι κάπως ατελές. Μην το θεωρείτε ότι είναι κάτι δεδομένο. δείτε από την εμπειρία μας. Είναι δυνατή και αντίστροφη κίνηση. Και αν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη βούλησή μα η σκοτία από την Ένωση, θα επιστρέψουμε. Και βασιζόμαστε σε εσά. Και τώρα λοιπόν για ένα λεπτό ο κύριος Μποκία. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλέ προκλήσει. Για να κερδιθούν οι προκλήσει πρέπει κανεί να είναι αξιόπιστο. Κυρία Φοντερ εσεί είπατε ότι θέλετε να αυξήσετε κατά 30% τι δαπάνε για την εξωτερική πολιτική, αλλά δεν αρκεί να το λέει κανεί αυτό για να μπορέσει να ξεπεράσει ε, τι διαφορετικέ θέσει που υπάρχουν από τα κράτη-μέλη. Ε, και διαρωτώ με ε, στα νησιά Φίτζη, στα Μπαρμπάντο, αυτά πραγματικά μα ενδιαφέρουν. Ο κύριο Τίμερμαν θέλει μια Ευρώπη που να είναι με την δώρα του για το κλίμα, αλλά αν οι τρίτε χώρε δεν κάνουν την δική του τη δουλειά, δεν υπερασπίζονται του δικού μα πολίτε και τι δικέ μα επιχειρήσει. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να υπάρχουν περισσότερα εργαλεία που θα εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορεί να αξιολογήσει αν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση είναι συμπαθητική ή όχι. Ε, θα μπορούσατε ίσω να σκεφτείτε να είσαστε μια επιτροπή χωρί αποκλεισμού, αλλά έχει έχετε απορρίψει την σύγκρουση με εκείνους τους ανθρώπους ε, που θέλουν ε, την εξέταση παρελθόντος. Καλή τύχη σας εύχομαι, γιατί πραγματικά την έχετε απόλυτη ανάγκη. Ο κύριος ε, Τσίλα για ένα λεπτό. Βρήκατε την ισορροπία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση τις ε, θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τις ε, κατανήματε πολύ καλά. Δύσκολο ήταν το καθήκον αυτό, αλλά μπορείτε και να βασιστείτε στην υποστήριξη πολλών ε, βουλευτών της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Αυτό θα ισχύει και το μέλλον, όταν δηλαδή η περιβαλλοντική πολιτική ε, δεν θα μπλοκάρεται. Ε, το ίδιο είπε πρόσφατα και ο πρώην πρόεδρος, αλλά μην ξεχνάτε, αν ακολουθήσετε την ίδια κατεύθυνση, θα έχουμε κάποια προβλήματα. Αν ε, υπονομεύσουμε την συνεργασία μας ε, ε, με τις ΗΠΑ και πάμε πιο ανατολικά, νομίζω ότι αυτό θα είναι αρκετά επικίνδυνο ως γεωπολιτική εξέλιξη. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Χάζεκα, παρακαλώ για ένα λεπτό. Αυτά που λέτε είναι εις βάρος των συμφερόντων των ανθρώπων και της φύσης. Αυτό το βλέπουμε με την ενεργειακή αλλαγή ή με τα ε, δηλητήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ μεγάλη δύναμη και είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ανεξάρτητη. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ξαφνικά να εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέροντα ε, σε πολυεθνικές εταιρείε όπως την Μονσάντο ή σε άλλες εταιρείε εξόριξης πετρελαίου. Μιλάμε για εκατομμύρια και θεωρώ ότι αυτό δεν θα επιτρέπει να υπάρχει μια σωστή πολιτική. Αλλά ακόμα και ο κύριος Τίμερμανς λέει ότι είναι απαραίτητο να γίνουν ε, κάποια πράγματα για να ε, αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, αλλά ε, είναι απογοητευτικό το ότι οι φιλοδοξίες της Επιτροπής δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν το δικό μας το κόμμα, το κόμμα των ζώων, δεν θα υπερψηφίσει την Επιτροπή. Για ένα λεπτό, κύριο Σίντσιτς. Ευχαριστώ πολύ. Παρουσιάσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πένους, παρουσιάσατε τους επιτρόπους, τα διάφορα χαρτοφυλάκια και είπατε ότι επιδιώκετε την αριστεία. Γι' αυτό και λοιπόν από πλευράς Κροατίας διαρωτώ με ε, γιατί επιλέξατε αυτή την επίτροπο από την Κροατία το κατεστημένο στην ε, Κροατία έχασε ένα εκατομμύριο πολίτες από την προσχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Σλαβωνία τα τελευταία έξι χρόνια χάσαμε κάθε τέταρτο μαθητή και φοιτητή. Ως εκ τούτου, κατά τη δική μου άποψη, δεν ε, έχει νόημα να επιλέξετε κάποιον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος δεν έχει ιδέα για τις ε, δημοκρατικές και δημογραφικές, με για τις δημογραφικές εξελίξεις. Βεβαίως ε, εσείς ε, στο Βερολίνο τα βλέπετε διαφορετικά. Εσείς απλά τώρα επιβραβεύσατε το κατεστημένο στην Κροατία και λέτε καλά να πάθουμε που χάσαμε τόσους πολλούς πολίτες. Αλλά αν συνεχίσετε έτσι, ξέρετε κάτι, τελικά στην Κροατία θα μείνουν μόνο συνταξιούχοι και πολιτικοί και όταν θα ανοίξει και η Αυστρία τις πόρτες της θα φύγουν και άλλοι. Ε, μια τέτοια χώρα πώς θα επιβιώσει, το έχετε σκεφτεί αυτό. 1,5 λεπτό κύριος Χαλίκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Βοντελάιν, εκ μέρου τη πολωνική αντιπροσωπεία στο ΕΛΚ και εκ μέρου τη πλειοψηφία τη πολωνική κοινωνία που είναι υπέρ τη Ευρώπη και τη Δημοκρατία, έχουμε μεγάλε ελπίδε για το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίδε για την ομάδα που μα παρουσιάσατε. Πράγματι, οι πολίτε ανησυχούν για την ποιότητα ζωή στην Ευρώπη. Γι' αυτό η πολιτική για το κλίμα και η προστασία του περιβάλλοντο είναι πολύ σημαντικά θέματα, αλλά και η υγεία η προστασία της είναι πολύ σημαντική. Με μεγάλη ικανοποίηση βρήκα ότι έχετε την υγεία σαν προτεραιότητα να καταπολεμήσετε αποτελεσματικά ε, το μεγαλύτερο φωνέα, το καρκίνο. Χρειάζεται συντονισμό για την εκτέλεση οικονομικών στόχων. Χρειαζόμαστε καλό προπολογισμό για κάτι τέτοιο. Θα ήθελαμε να είναι μεγαλύτερο, όχι μικρότερο ο προπολογισμό. Θα θέλαμε να έχουμε νέε θέσει εργασία που θα δημιουργηθούν. Εστιαστούμε επί τη καινοτομία και της ανάπτυξη τη οικονομία και τη ε, παιδεία. Υπάρχει κι άλλο θεμελιώδες θέμα που επανειλημμένα αναφέρατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων την προάσπιση της ελευθερίας των αξιών και του κράτους δικαίου είναι θεμελιώδες στοιχείο των κοινωνιών μας. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Όλες οι κυβερνήσεις είναι ίσες. Να είσαστε συνεπείς παρακαλώ στις δραστηριότητές σας, ούτω ώστε η κοινότητά μας να μην κινδυνεύσει και να μην υπονομεύεται από κανέναν. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχόμαστε καλή τύχη. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Τάνιτσεφ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε Επιτροπή. Σήμερα θα λάβετε μια ευρύτερη υποστήριξη και πιο παγιωμένη, έτσι, βέβαιη στήριξη από τους σοσιαλιστές από τον Ιούλιο. Και αυτό για τους εξής λόγους. Πρώτον, κύριε Πρόεδρε, δεσμευθήκατε σοβαρά ε, πολιτικά για προοδευτική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας αλλαγής που είναι κοινωνικής, κοινωνική, ε, οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσης. Η πιο προοδευτική πολιτική ατζέντα ε, είναι αυτή τη στιγμή επιτάπτως και εμείς οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Αλλά εμείς οι σοσιαλιστές θα είμαστε άγρυπνοι, απαιτητικοί για όσον αφορά την απόδοσή σας. Πρώτος σας είναι το PDP, διότι δεν μπορούν να ασκηθούν πολιτικές χωρίς πόρους. Έπειτα έχουμε μια ισχυρή ομάδα σοσιαλιστών επιτρόπων με όραμα, ε, αρμοδι... Ε, ικανότητες και ενέργεια. Και η Κομισιόν δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ως ε, έδρα του ΕΛΚ όπου ένα κόμμα κυριαρχεί στις πολιτικές. Είναι ισορροπημένο σώμα. Τρίτον, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν άλλη υπομονή. Θέλουν αποτελέσματα. Στις τελευταίες ευρωεκλογές υπήρξε συμμετοχή ρεκόρ, αλλά η υπομονή των πολιτών είναι στα όρια της. Οπότε παρακαλώ, αρχίστε να δουλεύετε και να αποδίδετε από σήμερα. Έχουμε μόνο πέντε χρόνια μπροστά μας. Για μισή λεπτό η κυρία Βόντεν. Sorry. Συγγνώμη, κυρία Βαντερ Λάιεν, Επίτροπε, Πρόεδρε. Ε, πήρε καιρό για να φτάσουμε εδώ και σήμαινε αυτό συμβιβαστικέ για πολλού. Όμω πλέον είναι και καινή ώρα η Ευρώπη να σταθεί στη δουλειά και να βγάλει πολιτικέ που να είναι ωφέλιμε για όλου του Ευρωπαίου. Κυρία Βαντελάιεν, θαυμάζω το τη, φιλοδο, τη φιλοδοξία σα για ισορροπία στα φύλλα. Λίγο σα μένει ακόμα, αλλά ποτέ δεν είχαμε τόσο έντονη γυναικεία εκπροσώπηση στι ανώτατε ηγετικέ θέσει τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ για αυτή σα δέσμευση. Και τώρα προσβλέπω σε παρόμοια ισορροπία σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ε, τόσο στις, ε, ε στις ε, χαμηλόβαθμες θέσεις όσο και στις υψηλόβαθμες και σε όλα τα θεσμικά όργανα. Βεβαίως, αντιπογοητεύτηκα που δεν υπάρχει Βρετανός Επίτροπος στην παρέα σας σήμερα. Ε, η ε, ανόητη μας κυβέρνηση έχει βλάψει την φήμη του έθνους μας. Θα σας διαβεβαιώσω όμως ότι όσοι έχουμε ακόμα τα λογικά μας θα δουλέψουμε για να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα και καλωσορίζουμε τη δική σας στήριξη. Στην Επιτροπή μας όταν σας υποδεχτήκαμε ως υποψήφια πρόεδρο είπατε ότι θα έρθετε σε επαφή με τους φιλοευρωπαίους Βρετανούς για τα γλωσσικά ζητήματα και για τα ζητήματα μετά ε, Brexit. Υπάρχουν ε, όμως λόγοι για αισιοδοξία. Εσείς σωστά ε, ιεραρχήσατε το κλίμα, την ψηφιοποίηση. Εγώ προσβλέπω στο να έρθω εδώ για έλεγχο κάθε θέμα με τη σειρά του, με πολιτικές που θα οδηγήσουν στην Ευρώπη σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι σήμερα. Κύριε Βαντελάιεν, είναι βαθιά μου επιθυμία να είμαι εδώ σε πέντε χρόνια για να δω τα αποτελέσματα της δουλειά την οποία ξεκινάτε σήμερα. Όπως είπατε, είναι φιλόδοξο και λαμπρό project και όλοι όλοι θα πρέπει να το τιμήσετε και να το εκτιμήσετε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ντελμπό Σκορφίλτ. ακόμα είναι νέα και εύθραστη η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, δεν έχει οριμάσει ακόμα και δεν είναι φεντεραλιστική. Τα κράτη-μέλη διορίζουν του επιτρόπου και αυτό επιτρέπει σε κυβερνήσει να στέλνουν επιτρόπου που του είναι πιστοί η Ουγγαρία και η Πολωνία. Και όμω το άρθρο 7 ήδη δρομολογήθηκε κατά αυτών των χωρών, διότι παραβίασαν το κράτο δικαίου και τι αξίε μα. Σήμερα, υποψήφοι που υποστάλλει από την Ουγγαρία θέλει να προσπέσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στι χώρε που θέλουν ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρόκληση για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε στα λόγια για το θέμα του κράτου δικαίου και για τι θεμελιώδει ελευθερίε. Θα είσαστε σε θέση πραγματικά να τα χειριστείτε αυτά παρά τι πιέσει των κρατών μελών και παρά τη μεγάλη ισχύ τη διαδικασία τη διακυβερνητική θα, είσαστε στη, στην, θα εκπηρετήσετε τι ευρωπαϊκέ αξίε και του πολίτε παρά να υπακούτε σε εντολέ των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε το ρόλο του απορρίπτοντα ε, τον υποψήφιου που είχαν συγκρούσει συμφερόντων και επίση και του υποψήφιου του άκουσε για την ανεξαρτησία του και τι ικανότητε που έχουν με τη σειρά σα να είσαστε εσεί γενναία. Το χαρτοφυλάκιό σα δεν άλλαξε. Ένα χαρτοφυλάκιο δεν άλλαξε τίτλο. Ονομάζεται Δημοκρατία και Δημογραφία. Για μια φεμινίστρια αυτό με κάνει να τριχιάζω αυτό ο τίτλο. Και η επίτροπο η κυρία Σουίτσα είναι επιφορτισμένη με τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Κατά να ακούσει τη αυτή υποψήφια αρνήθηκε να καταδικάσει τη θεωρία τη μεγάλη την κατάσταση. Ή ακόμη φορά βλέπετε ε, ανησυχούμε μπορείτε να διαβολήσετε ε, να έχουμε ένα μέλλον στην Ευρώπη που θα προστατεύει τι θεμελιώδει ε, αρχέ και το φεμινισμό Κυρία μου, υπάρχει γαλάζια κάρτα για σας. Κυρία Ντελμπός, κυρία Ντελμπός, ο κύριος Ότος έχει σηκώσει γαλάζια κάρτα. Δέχεστε την ερώτησή του. Είπατε ναι ή ου. Ναι. Όχι. Με μπερδέψατε. Δέχεστε τη γαλάζια κάρτα. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι. Ναι. Ωραία. Κύριε Ότος, έχετε το λόγο. Okay, Ας προχωρήσουμε. Ας τα αφήσουμε αυτό, ας προχωρήσουμε. Έτσι. Ευχαριστώ για τον γέλο, τα βοηθά. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Κρά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, λαμβάνουμε υπόψη μας ότι αυτή η Επιτροπή πράγματι ακολουθεί μια ημερήσια διάταξη ε, αριστερή ε, βέβαια αυτό εντυπωσιάζει, γιατί τα αποτελέσματα των εκλογών έδειξαν ότι οι πολίτες θέλουν περισσότερο συντηρητική κατεύθυνση. Ως βασικό σας θέμα επιλέξατε το κλίμα, το αν θα μειωθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κατά ένα ή δύο βαθμούς, αλλά ξέρετε δεν είναι αυτό βασικά που απασχολεί τους ανθρώπους. Ανησυχούν για τη μετανάστευση, για τη δουλειά τους, αν είναι εξασφαλισμένες οι θέσεις τους, το μέλλον της πατρίδας τους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η Επιτροπή ε, πράγματι ακολουθεί αυτά τα οποία οι περισσότεροι θεωρούν σημαντικά, όμως ε, δυστυχώς ε, δεν είναι αυτά τα οποία επιτιμούν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα σας παρακολουθούμε με κριτικό πνεύμα και θέλω να σας πω ότι εμείς δεν θέλουμε ιερείς ε, αριστερής θρησκείας, θέλουμε εκείνους που θέλουν το κοινό καλό και φοβούμεθα ότι αυτό δεν θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Έπινγκ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, το Green Deal, το Πράσινο Σύμφωνο, είναι το μεγάλο εγχείρημα αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα είμαστε ουδέτεροι απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ως προς το αποτύπωμα κυρίως, αλλά δεν άκουσα πώς θα γίνει αυτό. Εγώ έχω διαβάσει όλα τα έγγραφα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μερικοί τα αντιμετωπίζουν αυτά τα έγγραφα ως τη βίβλο. Λένε ότι μέχρι και 500.000 ευρώ ε, το χρόνο αυτό θα κοστίσει για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και μετά πιο κάτω λέει ότι σε 20 χρόνια ε, θα έχουμε φτάσει σε 11,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή τριπλάσιο το ποσό από το ΑΕΠ της Γερμανίας. Ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το ΑΕΠ της Γερμανίας. Γι' αυτό λοιπόν έχω μία πολύ απλή ερώτηση κύριε και κύριοι. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Ποιος θα τα πληρώσει και όταν την έκανα την ερώτηση δεν άκουσα απάντηση να σας πω ποιος θα τα πληρώσει. Οι φορολογούμενοι. Αυτοί θα τα πληρώσουν. Αυτοί ε, θα έχουν υψηλότερους λογαριασμούς ε, ρεύματος. Αυτοί θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και ήδη στην Ολλανδία βλέπω ότι γίνονται μικρές εξεγέρσεις. Εξε, εξεγείρονται οι οικοδόμοι, οι εργάτες γιατί δεν μπορούν πια να πληρώσουν. Άρα δηλαδή πολλά έχετε να δουν, πολλά έχουν να δουν τα μάτια σας. Κύριε Επίνκ, υπάρχει μία μπλε κάρτα από τον κύριο Κόκαλη. Δέχεστε την μπλε κάρτα του κύριου Κόκαλη. Βεβαίως, τη δέχομαι. Παρακαλώ κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο. 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Έπικα, αναφερθήκατε στο κόστος ε, της, του νέου πράσινου συμφώνου μέχρι το 2050 και θέλω να σας πω ότι οι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι μέχρι το 2050 αν δεν γίνει τίποτα θα φτάσουμε σε κόστος 3 εκατομμύρια. Έχετε λοιπόν υπόψη σας το πόσο θα κοστίσει τελικά το να μην κάνουμε απολύτως τίποτα σχετικά με το κλίμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, το καλύτερο θα ήταν να τροποποιηθεί το πράσινο σύμφωνο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουμε στην πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον. Γνωρίζω ότι πολλά κοινοβούλια δεν συμφωνούν. Είναι όμως σημαντική η πυρηνική ενέργεια και πρέπει να διατηρήσουμε και το φυσικό αέριο. Στην Ολλανδία πρόκειται να καταργηθεί το φυσικό αέριο. Κακό αυτό γιατί κοστίζει, κοστίζει πολύ. Το φυσικό αέριο είναι φιλικό θετικό προς το περιβάλλον. Επίσης, τη βιομάζα, να μην τη χρησιμοποιούμε πια. Η βιομάζα δεν είναι πράσινη, όπως ισχυρίζονται οι πράσινοι. Δυστυχώς, ο μιλητής διακόπτεται. Για ένα λεπτό, κύριο Σαρβανίτης, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, είχατε πραγματικά μια εξαιρετική σκηνική παρουσία. Υποσχεθήκατε τα πάντα στους πάντες, μάλλον όχι στους πάντες, αλλά σε συγκεκριμένα συμφέροντα και σε συγκεκριμένε πολιτικές απόψεις μας είπατε για στρατικοποίηση της ευρώπης για το περιβάλλον έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη για εσάς δεν μίλησατε καθόλου για τα εργατικά δικαιώματα για τη διαφθορά και τη διαπλοκή δεν μας πείσατε για το προσφυγικό επιμένετε στον απαράδεκτο για μας τίτλο προστασία ή πρόθεση ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. δεν ακούσατε καθόλου καμία πολιτική ομάδα εκτός από το ε, κόμμα σας δηλαδή όπως είπε ο κύριος Βέμπερ έχει το λαϊκό κόμμα πρόεδρο στην κομισιόν. δεν είναι έτσι. χρειάζεται σύνθεση και με τη σύνθεση δεν τα πάτε και πολύ καλά από ό,τι φαίνεται από την αρχή οπότε θα πάμε στο άλλο επίπεδο της δημοκρατίας που είναι η πολιτική σύγκρουση. καλό κουράγιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βοντελάιν, μετά από δύσκολες παρατεταμένες εργασίες για να ετοιμάσετε την Ευρωπαϊκή σας Επιτροπή και το αρνητικό μήνυμα που παρατήσατε το σύστημα τη Πίτσα Καντιτάτ για την εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να είστε ικανοποιημένοι και σας συγχαίρουμε που ετοιμάσετε μια ομάδα επιτρόπων, ένα σώμα και τους βάλατε πίσω από ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Για να είσαστε επιτυχείς στο τέλος της θητείας σας, πιστεύω ότι θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Ε, καταρχάς, πιστεύω ότι πρέπει να ξανακερδίσετε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, ενισχύοντας ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι θα ήταν μια καλή αρχή να διερευνήσετε κάποιες από τις προτάσεις του κυρίου Βέμπερ ε, αυτό που ανέφερε στο πολίτικο χτε στη συνέντευξή του. Το δεύτερο είναι πολιτική και δράση. Ο κοινωνικό ε, πυλώνα πρέπει να ισχυθεί όχι μόνο το ελάχιστο εισόδημα, αλλά και οι διαφορέ αμοιβών θα πρέπει να μειωθούν στην Ευρώπη και να εξαλειφθούν. Η αλλαγή του κλίματο για το κάτω δικαίου χρειάζονται ενέργεια και θα πρέπει να δώσετε απαντήσει σε αυτά τα θέματα για να αντιταχθείτε στα επιχειρήματα και σε επικρίσει των λαϊκιστών και των ευρωσκεπτικιστών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Να κάνω μια ανακοίνωση. Έχουμε 15 ανθρώπους που ζητούν να μιλήσουν στο Catch the Eye και για να είμαι δίκαιη έναντι εκείνων που θέλουν να προσθεθούν στη λίστα, πρέπει να πω ότι πρέπει να κλείσει τώρα ο κατάλογο, διότι κάποιοι θα απογοητευτούν. Και τώρα για 1,5 λεπτό δίνω το λόγο στον κύριο Μούρεσαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε Βοντελάιν, καλώ ήρθατε ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη σημερινή ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι είμαστε ενωμένοι από το καθήκον που έχουμε να δώσουμε τι καλύτερε πολιτικέ για του λαού τη Ευρώπη. Μπορεί να διαφωνούμε όσον αφορά ε, τι λεπτομέρειε, αλλά αυτό είναι το κοινό καθήκον για μα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα από τα βασικά εργαλεία στη διάθεσή μα για να δώσουμε αποτελέσματα είναι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα 7 χρόνια. Και πρόεδρο Βοντελάια, να σα πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι περιμένει από αυτόν τον τομέα. Όλοι είδαμε του λαού τη Ευρώπη να ψηφίζουν. Φοιτητέ, γεωργοί, μικρομεσαίε επιχειρήσει, κόσμο που περιμένει περισσότερο για την ασφάλεια, περιμένουν να έχουμε αποτελέσματα για την αντιμετώπιση αλλαγή του κλίματο και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί έναντι των λαών τη Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με πολύ λιγότερα. Αν συμφωνούμε συμφωνούμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει περισσότερο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σαφή. Νέε προτεραιότητε απαιτούν και χρηματοδότηση. Παρακαλώ να έρθετε στάξει μα μαζί, κυρία Βοντελάη, να πείσετε τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να δώσουν τελικά χρήματα για να ελοπίσουν αυτά που λένε στι δηλώσει. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο τομέα. Πού πρέπει να επενδύσουμε. Πρέπει να βρούμε ισορροπία μεταξύ παλαιών και νέων προτεραιοτήτων. Συνοχή, γεωργία, μόνο επειδή ήταν προτεραιότητες επί δεκαετίες, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ξεπερασμένε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε εκεί, αλλά βεβαίω πρέπει να επενδύουμε και στο ψηφιακό ε, κλάδο, το κλίμα κλπ. Και μετά για το χρονισμό. Σημαντικό ο προπολογισμό, αλλά είναι κάτι που χρειάζεται κατεπηγόντω επίση να συνεργαστούμε, ώστε το Δεκέμβρη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πετύχουμε μια κοινή συνεννόηση περί των προσδοκομένων από την Ευρώπη και τι περιμένουμε τον προπολογισμό. Α μην ξεκινήσουμε με μικροσυζητήσει για στοιχεία και αριθμού, διότι θα είναι κάτι διχαστικό. Η πολιτική συμφωνία για τα προσδοκόμενα πρώτα απ' όλα και μετά τελικά να δώσουμε τα χρήματα για να ελοποιηθούν οι προσδοκίε και οι υποσχέσει μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σα. Κυρία Ντάλη, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα το πρωί μιλάμε με μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει δεσμευτεί να βάλει το πράσινο σύμφωνο στην προτεραιότητα. Το πράσινο σύμφωνο θα παραμένει, πρέπει να παραμείνει λόγος και τίτλος, να γίνει πραγματικότητα που θα κάνει θετική διαφορά για τη ζωή των πολιτών, όπου και να ζουν αυτοί, ανεξάρτητα από το μέγεθο τη χώρα του. Ξεκινώντας λοιπόν μια ένα σοβαρό πρόγραμμα, εφαρμογή πρόγραμμα για την απαλλαγή από το άνθρακα που στο επίκεντρο θα έχει τη μεταποίηση, την αλλαγή τη βιομηχανία, τον ισχύ στην ανταγωνιστικότητα και το πράσινο σύμφωνο θα πρέπει να ξεπεράσει του απλού στόχου, να είναι μια επανάσταση για την επιχειρηματικότητα και για τι βιομηχανίε μα. Θα πρέπει να έχουμε μια επανάσταση στον τρόπο που κινούμε, θα δρούμε και βοηθούμε του εργαζόμενου να αποκτήσουν νέε δεξιότητε και πώ να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μα για τι μελλοντικέ βιομηχανίε. Έχουμε βιομηχανίε και επιχειρήσει οι οποίε καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται αυτή η μεταμόρφωση και η μετάβαση και βλέπουν τους θεσμούς για σαφείς δεσμεύσεις. Και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες το πράσινο σύμφωνο είναι μια νέα δυνατότητα να εξασφαλίσουμε ένα νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο τους εργαζόμενους και τους πλέον ευάλωτους τους βάζει στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Είναι μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με γειτονικές υπήρους όπως είναι η Αφρική παραδείγματο χάρη, να προωθήσουμε συνεργασίες και να δώσουμε σαφέστερη ανανεώσιμη ενέργεια και είναι η δική μας ευκαιρία να προστατεύσουμε την κοινωνική ευημερία όλων των πολιτών μας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπουμε στο να είμαστε εταίροι σε αυτή τη μετάβαση, στη μεταμόρφωση για να δείξουμε σαφώ στου πολίτε μα, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, ότι το εγχείρημα το ευρωπαϊκό ζει και δίνει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. For and Για 1,5 λεπτό, κύριο Ασμάνη. ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Ορισμένες εξ αυτών είναι απειλές, αλλά άλλες είναι ευκαιρίες. Δεν μπορούμε να σταθούμε άπρακτοι ε, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Πρέπει να ανανεωθεί η Ευρώπη Το ρεκόρ συμμετοχή στι τελευταίε ευρωεκλογέ πριν από έξι μήνε μα δείχνει πω οι Ευρωπαίοι πολίτε μα εμπιστεύονται. Όμω σε αντάλλαγμα αναμένουν να του προσφέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, ε, γι' αυτό και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει τη δουλειά όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε να μπορέσουμε να αποδίδουμε στις υποσχέσεις μας για μια Ευρώπη ισχυρότερη που δουλεύει για τους λαούς μας. Το, αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι λίγο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να εξασφαλίσουμε μια σταθερή οικονομία, να καινοτομήσουμε, να αντιμετωπίσουμε την ε, ψηφιακή ατζέντα, αλλά και να ελέγξουμε τα πράγματα, να ελέγξουμε ελέγξουμε τη μετανάστευση και να παρέχουμε ασφάλεια και σταθερότητα σε έναν μη σταθερό κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε επίσης πάντα στους παλιούς μας σύμμαχους. Γι' αυτό και η νέα Επιτροπή ε, την παροτρύνω να αρχίσει να συνεργάζεται με, το, με τη νέα Ευρώπη ώστε να έχουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για μια ευημερή Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Είμαι ευτυχής που σας βλέπω κυρία Πρόεδρε και ελπίζω πως μαζί θα αρχίσουμε τη δουλειά για μια ανανεωμένη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Εκχάουτ για ένα λεπτό τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ε, σας ευχαριστώ πολύ για τις προτεραιότητές σας που ακούγονται σωστές και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για αυτές. Αλλά είναι επίσης σαφές πως έχουμε τις δικές μας ανησυχίες που έχουν ε, αναφερθεί και παλιότερα από τη Αλέρα. Αφορούν το κράτος δικαίου, την κοινωνική διάσταση της εσωτερικής μας αγοράς, αλλά και την ανθρώπινη μεταχείριση, αντιμετώπιση των προσβήγων εντός και εκτός Ένωσης. Υπάρχουν ανησυχίες λοιπόν και γι' αυτό δεν θα σας δώσουμε λευκή επιταγή, αλλά θα συνεργαστούμε μαζί σας για το Πράσινο Σύμφωνο για την ψηφιοποίηση στην εξασφάλιση ότι αυτές οι επικοινωνίες και για την Πράσινο Σύμφωνο που περιμένουμε σε δύο εβδομάδες ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα πέρα από τα ωραία λόγια ε, όταν πρόκειται για νομοθεσία ώστε να αλλάξουμε πραγματικά τον τρόπο ζωής μας μέσα στα πλανητικά μας σύνορα. Ε, γι' αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθήσει η Ευρώπη και θα δουλέψουμε για τις πραγματικές νομοθεσίες που θα έρθουν αργότερα και εκεί περιμένουμε πραγματική δράση. Ας πούμε, κλιματική νομοθεσία επόμενη χρονιά θα είναι η μόνη και τελευταία ευκαιρία ώστε οι φιλοδοξίες μας να είναι ψηλότερες πριν να ξεκινήσει πραγματικά το Παρίσι. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την στιγμή αυτή και θα συνεργαστούμε μαζί σας ε, για αυτό το σκοπό. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, η κυρία Φοντερ Λάιν πράγματι πέτυχε να συγκεντρώσει εδώ την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως μερικές φορές ε, να την εντύπωση μιας άχρωμης ε, Επιτροπή, αλλά δεν είναι αλήθεια. Η κυρία Φόντερ ενδιαφέρεται περισσότερο για αριστερά εγχειρήματα και προγράμματα τα οποία βοηθούν την πολυμέρεια. Η κυρία Φόντερ θα πρέπει λοιπόν να ε, τραβήξει τα σχοινιά ε, και να ε, προάγει περισσότερο τον φεντεραλισμό στην Ευρώπη. Αυτό όμως είναι σε αντίφαση με την ελευθερία των ευρωπαϊκών λαών. Η Φλάνδρα, μελλοντικό κράτος φλάνδρα, να ξέρετε, θα σας καταδείξει το δρόμο. Για ένα λεπτό η κυρία Κάνκο. Α, η διεύρυνση μας έχει δείξει ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής ε, είναι κάτω Και Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλέ απειλέ στη διαχείριση των συνόρων, Κυρίω από πλευρά Τουρκία α μην κλείνουμε τα μάτια, πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσει. Όλοι θέλουμε η Επιτροπή να παρουσιάσει αποτελέσματα και γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να ενώσετε την κατακαιρματισμένη Ευρώπη, να επιτύχετε πλειοψηφίε για ένα σημαντικό θέμα που είναι κυρίω ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Να υπάρχουν αποτελεσματικέ λύσει σε θέματα εσωτερική ασφάλεια διαχείριση τη μετανάστευση και οικονομία στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και εκεί πρέπει να υπάρχει προστασία. Στο εμπόριο να προστατεύουμε το περιβάλλον μας ενώ θα διασφαλίζουμε ότι η Ευρώπη θα παραμένει ανταγωνιστική. Αυτό δεν είναι αμεληταίο εγχείρημα αλλά είναι ε, σημαντικό. Η Σουφραζέτα παλαιότερα ε, είχε πει, μια γνωστή Σουφραζέτα είχε πει ότι η Ευρώπη και ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα δικείται από γυναίκες. Εσείς είσαστε η ελπίδα για μας ε, και προσβλέπω στο να συνεργαστώ μαζί σας. ένα λεπτό, Κυρία Βαντελάιεν, αυτή η Επιτροπή δεν απαντά σε ούτε ένα από τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι είναι το χειρότερο δεν αλλάζει και όσα αλλάζουν, αλλάζουν προς το χειρότερο. Η μόνη γλώσσα της Επιτροπής για την Πολιτική Οικονομία είναι η λιτότητα και η επιλογή για τον Αντιπρόεδρο της, για την, υπεύθυνο για την οικονομία ακριβώς δείχνει τη συνέχεια σε αυτή την λιτότητα και την, όλες οι πολιτικές που μας εκφράσατε που μπορεί να ξεπεράσουν ε, την λιτότητα υποτιμούνται. Ας πούμε, η πολιτική συνοχή ε, ε, υπόκειται φοβερή περικοπή. Η πράσινη, το Πράσινο Σύμφωνο έχει έναν αντιπρόεδρο που προχωρά σε δημόσιους δηλώσεις και ζητώντας πόρους για τις πολιτικές τους. Πολιτικές τις οποίες δεν μας έχει ακόμα παρουσιάσει. Ε, ε, πρόκειται για ε, πολλά λόγια και λίγα αποτελέσματα. Δηλαδή ένα μικρό δημοσιονομικό φάκελο για πολιτικές τις οποίες δεν πρόκειται να μπορέσει να επιβάλλει η Επιτροπή και γιατί η πλειοψηφία εδώ προτιμά πολιτικό μπλοκάρισμα 5 ετών από ότι ένα θεσμικό μπλοκάρισμα κάποιων μηνών. Καμία φιλοδοξία Τίποτα δεν μπορεί να κινητοποιήσει αυτό εδώ το σώμα ε, υπέρ αυτής της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ την πρόεδρο της Επιτροπής που λέει ότι, θέλει να ότι είναι Remainer, η διευκρίνηση είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Να πω ότι είναι καταστροφική αποκάλυψη και τελικά ε, εκεί χάθηκε το θέμα του Brexit προειδοποίηση ότι θα κινηθεί νομικά κατά τη χώρα μου η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αρνηθήκαν προτείνουμε ε, επίτροπο. Αλλά τι νόημα έχει, φεύγουμε ούτω ή άλλω. Και αυτόν που είχαμε, ο Κίνο και Μάντελσον, αυτοί ε, χρησιμοποίησαν αυτό σαν ε, ευκαιρία για να μαζέψουν χρήμα, 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι φεντεραλιστές και δεν μπορούν να προστατεύσουν τους λαούς τους, απλώς θέλουν να συμμορφώνονται και να μαζεύουν λεφτά. Οπότε δεν μας δεν ασχολούμαστε καν. Η απόφαση της χώρας μου που επιβεβαιώνει ότι πράγματι φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. And remember. Και θυμηθείτε, εάν σας δημιουργούμε πολλά προβλήματα, μπορείτε πάντα πρώιμα να μας δώσετε μια κλωτσιά να μας διώξετε. Um, um Harris. Κυρία Χάρη, δύο πράγματα. Ίσως να σε εκπλήσει αυτό. Εγώ είμαι Remainer επίσης, θέλω να παραμείνω το Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεύτερον, δέχεστε γαλάζια κάρτα του κυρίου Σμιθ. Κύριε Σμιθ, για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Χάρης που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω. Είναι νομική υποχρέωση διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτο δικαίου και δικαιοσύνη. Θα πρέπει να διορίσει επίτροπο ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, το παραβιάζει, γιατί έχουμε μια ανεύθυνη κυβέρνηση, μηδενιστική εμείς έχουμε προνόμια σαν ευρωβουλευτές. Είσαστε υπέρ να παραιτηθείτε εσείς από το μισθό σας και τα επιδόματά σας για το χρόνο που είσαστε εδώ, αν είσαστε ε, ικανοποιημένοι να αποχωρήσετε. Under UK law we also can't... Σύμφωνα με τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια προκλητικής ε, περίοδου. Και δεύτερον, Επίσης πρέπει να λογοδοτήσουμε στο λαό της Βρετανίας. Δεν λογοδοτούμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το καταστήσαμε σαφέστα το 2016 όταν ψηφίσαμε να αποχωρήσουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, Κυρία μου. Και σε ευχαριστώ παρόλα αυτά για 1,5 λεπτό. Η κυρία Μονσεράτ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, ε, Πρόεδρε Βαντερ Λάιεν, σα ζητάμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο ενωμένη και πιο ασφαλή. Ισχυρή για να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει θέσεις απασχόληση. Ενωμένη ώστε τα κράτη δικαίου να αντιμετωπίσουν του Εθνικισμού και του λαϊκισμούς που τα απειλούν. Και ασφαλή για να μπορέσει να υπερασπιστεί τα εξωτερικά μα σύνορα, να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και να υπερασπιστεί τι δημοκρατίες ανά τον κόσμο. Επίση Επίσης χρειαζόμαστε μια Ευρώπη πιο χρήσιμη για όλους τους Ευρωπαίους. Να είστε χρήσιμοι ώστε οι νέοι να έχουν ευκαιρίες, ώστε οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, γιατί η απασχόληση είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική για να μην μείνει κανείς πίσω. Εμείς θέλουμε να έχουμε μετανάστευση νόμιμη και να είμαστε χρήσιμοι για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφική πρόκληση της γυραιάς μα Υπήρου, να φροντίσουμε τον κόσμο της να υπερασπιστούμε την υγειοργία μα, την κτηνοτροφία μα και την αλληλεία μα. Να συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών για να φροντίσουμε τον πλανήτη μα. Και κυρίω πρέπει να ηγηθούμε τη τεχνολογική επανάσταση, τη καινοτομία και τη ψηφιοποίηση. Να είμαστε χρήσιμοι και πιο κοντά στου πολίτε μα, να φτιάξουμε την Ευρώπη των ανθρώπων και τη ισότητα. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη με πιο ε, ε μεγαλύτερη εγκύτητα στου πολίτε, μεγαλύτερη δημοκρατία, έτσι μόνο θα επιτύχουμε σε αυτό το χώρο ειρήνης, ισότητας και ανάπτυξης. Είμαι βέβαιη ότι η Πρόεδρος θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έχετε την πλήρη στήριξη του, του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος. Για 1,5 λεπτό η κυρία Πύρη. Κυρία Πρόεδρε, είχαμε ε, την, τον αγώνα πριν από τις εκλογές για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Φοβάμαι ότι τελικά δεν τα καταφέραμε.